Καλημέρα σας. Έχουμε μία ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 6 δεν είναι κανεί ο οποίος θα είναι παρόν. Πρόκειται για τη μία ημερήσια διάταξη για τις νέες ε, δεξιότητες και προσόντα. Οπότε αυτό θα πάει στην επόμενη συνεδρίασή μας. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη. Σήμερα Έχουμε τα πάντα εκτός από εστονικά, λετονικά, λέει προ... ε, λιθα, λιθουανικά, μαλτέζικα, τσέχικα και σουηδικά. Όλες οι άλλες γλώσσες παίζουν και προς και από. Σημείο 3 ημερησίες διάταξης. Μαζί μας σήμερα έχουμε την Γενική Συγγήτρια για το 2012 <coughs> την κυρία Μπαλτσάνη, Φραντσέσκα Μπαλτσάνη, <coughs> η οποία θα μας παρουσιάσει τις απόψεις για το επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012. <coughs> Αλλά η κυρία Λοχμπίλντερ δεν είναι ακόμα παρούσα που είναι η συγγήτριά μας. Θα ακούσουμε λοιπόν καταρχήν αυτά τα οποία έχει να μας παρουσιάσει η κυρία Μπαλτσάνη. Σας παρακαλώ να ξεκινήσετε κυρία Μπαλτσάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συναντηθώ μαζί σας. Η διαδικασία του προπολογισμού βρίσκεται στην απαρχή της ακόμα, αλλά αυτή η απαρχή είναι μια ιδιαίτερα λεπτή χρονική στιγμή. Γιατί θα πρέπει να κατανοήσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα όλη την εργασία που θα πρέπει να αναπτύξουμε τους επόμενους μήνες. Όπως είδαμε πέρσι με μία μονάχα ανάγνωση του προϋπολογισμού και μία νέα μορφή ισότητας και ισοδυναμίας των ε, θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου δηλαδή και του Κοινοβουλίου, τα πράγματα απεδείχθησαν αρκετά λεπτά και ευαίσθητα. Και ιδίως λόγω των ε, αδιαφυσβήτων δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες πιέσεις προς την κατεύθυνση κα... περικοπών και περιστολών, πολλές φορές ακόμα και αδικαιολογήτων. Η άποψή μου, επομένω, ήταν από την αρχή η εξή, μια άποψη που την έχουν υποστηρίξει οι συνάδελφοι της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών που με έχουν υποστηρίξει με γενναιόδερο τρόπο. Ο στόχος μου ήταν να εμπλέξουμε στο βαθμό του δυνατού, ώστε γίνεται περισσότερο, τις επιμέρους επιτροπές γιατί ο προπολογισμό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, όχι μόνο στη μορφή αλλά και στο περιεχόμενο. Είναι η μόνη διαδικασία όπου είναι απαραίτητο από την αρχή όλοι οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν με τρόπο ενεργά. Και διότι ως συμμετέχοντες σε ειδικευμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστό προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιες θέλουμε να είναι οι προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού του 2012. Για το 2012 λοιπόν η πρότασή μου <clears throat> είναι καταρχήν να καθορίσουμε προοπτικές οποίες και προτεραιότητες οι οποίες θα εγγράφονται πλήρως στη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Επομένως, η κάθε επιτροπή θα πρέπει να δει ποιε είναι οι πιο λειτουργικές προτεραιότητες ως προς την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Όπως ξέρετε, η στρατηγική 2020 είναι μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, αλλά είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από τώρα να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας, εάν φυσικά θέλουμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ένα οδικό χάρτη ο οποίος θα μας βοηθήσει στην υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης στρατηγικής. Επομένως, το σημείο αναφοράς και η, ο βασικός άξονας αυτής της διαδικασίας είναι οι λεγόμενες πρωτοβουλίες φάρη, οι οποίοι θα πρέπει να καθοδηγούν την, ε, την Επιτροπή μας. Έχουμε παραγωγή χάρη να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στον σχολικό πληθυσμό της Ευρώπης που υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν τελειώνει το σχολείο και η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει φτάσει σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση για να μπορέσει να αναπτύξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεδομένου ότι οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας δείχνουν ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για εργασία με υψηλά προσόντα. Δυστυχώς ακόμα στην Ευρώπη εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη ανισότητα σε ό,τι αφορά την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων όταν συγκριθούμε με άλλες σημαντικές οικονομίες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλαίσιο λοιπόν της στρατηγικής Ευρώπη 2020 δίνει σημαντικά σημαντικές ε, αρμοδιότητες στην Επιτροπή σας για την ανάπτυξη ορισμένων αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα είναι αρμοδιότητες οι οποίες θα καθορίσουν την επιτυχία. Ε, φυσικά οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περιορισμένα κονδύλια Προτού συζητήσουμε για το τι θα γίνει για το τελευταίο έτος προγραμματισμού το 2013, ξέρουμε ότι και για το 2012 τα πράγματα είναι ήδη αρκετά στενά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν για το καθορισμό των προτεραιοτήτων τις οποίες θα θέλουμε να θεσπίσουμε, να συντονίσουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας και να έχουμε μια συγκροτημένη δημοσιονομική προσέγγιση για προοπτικές τις οποίες θεωρούμε πραγματικά χρήσιμες. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το πακέτο των πιλωτικών δράσεων και προπαρασκευαστικών εργασιών. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συγκρότηση αυτού του πακέτου, διότι η χρήση των πόρων για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά σχέδια καταλαμβάνει ένα τμήμα του περιθωρίου του προπολογισμού και επομένω μας μειώνει στη συνέχεια το περιθώριο ελιγμών. Πρόκειται λοιπόν για δράσεις, πολλές από οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και χρειάζεται επομένως να υπάρξει μεγάλη προσοχή για το πώς θα επιλέξουμε αυτές τις δράσεις, να εξετάσουμε κατά πόσο έχουν λειτουργήσει σωστά, να αξίζει τον κόπο να συνεχιστούν ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για άλλους σκοπούς. Ούτως, η πρώτη μας αυτή επαφή θα έχει σαν στόχο να σημαδεύσει την αρχή μιας διαδικασίας που ελπίζω θα συνεχιστεί με τη δική σας πλήρως εμπλοκή ως ειδικευμένης επιτροπής για τα θέματα του προϋπολογισμού. Με το πρώτο βήμα αυτό του καθορισμού των προτεραιοτήτων που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά το σχέδιο προϋπολογισμών που θα παρουσιάσει η Κομισιόν στις 20 Απριλίου και στη συνέχεια να έχουμε την καλύτερη ικανότητα να παρουσιάσουμε μια δική μας κοινοβουλευτική θέση καταθέτοντας τροπολογίες σε σχέση με το σχέδιο αυτό προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε πως η Επιτροπή σκοπεύει να καταθέσει σχέδιο προϋπολογισμού στα τέλη Απριλίου. Μια ανάγνωση μόνο θα έχουν ουσιαστικά το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο και θα δούμε αν χρειαστεί μια ούτως επίν άτυπη διαδικασία συνδιαλλαγής να μεσολαβήσει για να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παλτσάνη που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό και η προκάτοχό σα έκανε το ίδιο, αλλά στο παρελθόν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν ορισμένες φορές επιλογές στον προϋπολογισμό οι οποίες ήταν μάλλον αμφίβολης αξίας και με την κυρία Τρίπελ είχαμε επιμείνει ιδιαίτερα στο αντιμετωπίσουμε αυτό. Ε, θα έλεγα να δώσουμε στον κύριο ε, την ε, το λόγο για να μας πει τι βλέπει από το τελευταίο χρόνο για τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σε αυτή τη συνεδρία, κυρία Μπαλζάνη. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε στο εκπαιδευτικό θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι ε, αναρωτιόμουν πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση, διότι ο νέος τρόπος μεθόδευσης με όλες τις ερωτήσεις και τα ερωτήματα αναρωτιόμουν αν θα τα καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν ε, περιμένετε να σας δώσουμε ήδη τις προτεραιότητές μας. Δεν είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να συναντηθούμε ή να συνεδριάσουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Βεβαίως, άτυπα μπορούμε να ξαναβρεθούμε με τα γενέστερα, ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε. Θα ήθελα να σας πω πώς κατά τη γνώμη μου μπορείτε να συμβάλλετε και τι είδους προτεραιότητες θα πρέπει νομίζω να προσδιορίσουμε. Όπως, και, όπως είπατε κι εσείς, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβάλλει περισσότερο στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Συμφωνούμε με αυτό σε αυτή την Επιτροπή και ήδη πέρυσι ε, καταφέραμε να πετύχουμε κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε όμως έλλειψη χρηματοδότηση για τη στρατηγική περσέ και ήταν κάπως αρνητική έκπληξη για μας το Κοινοβούλιο η διαπίστωση αυτή κατά την άποψή μου δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο όπως το 2011. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη στρατηγική για το έτος 2020. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα τα οποία πρώτα απ' όλα θα προωθήσουν την κοινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, που θα βελτιώσουν τα προσόντα μας, την ανταγωνιστικότητα βεβαίω και θα διατηρήσουν την εξάπλωση της ε, κοινωνίας των γνώσεων. Βεβαίως επενδύουμε σε ανθρώπους. Αυτός είναι ο βασικός μας πρωταρχικός στο σκοπός εδώ. Έχουμε δύο προγράμματα ε, ε, που ασχολούνται με τους ανθρώπους. Το ένα είναι το πιο γνωστό στους νεότερους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Lifelong Learning, μέσα στο πλαίσιο δηλαδή της διαβίου και πρόκειται για το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο είναι τεράστια επιτυχία. Ε, είναι πετυχημένο πρώτα απ' όλα γιατί έχει μεγάλη απορροφητικότητα 100% περίπου για το Εράσμους και οι φοιτητές και ερευνητέ βελτιώνουν τα προσόντα τους, τις δεξιότητές τους ε, με αυτά τα προγράμματα, κυρίως δε τις γλωσσικές τους ικανότητες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε άλλους πολιτισμούς και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους. Και ακριβώς θα ήθελα να ενισχυθούν τα κονδύλια για τη διαβίου μάθηση. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω που μας ενδιαφέρει είναι το πρόγραμμα SPOTS. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε πρόγραμμα αυτού του τύπου μέχρι τώρα. Θα θέλαμε να είχαμε ένα. Τουλάχιστον θα θέλαμε να έχουμε κάποια καντήλια για να τα αναπτύξουμε. Ε, δεν μας δόθηκε σχεδόν τίποτα πέρυσι και νομίζω ότι αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι αυτά τα προγράμματα για σπορ ε, πρέπει να αναπτυχθούν, πρέπει τουλάχιστον να αποκτήσουμε ένα. Θα σταματήσω σε αυτό το σημείο, ανέφερα δύο-τρία σημεία που μας ενδιαφέρουν. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί θα προσθέσουν κι άλλα. Ε, σας έδωσα τις πρώτες μου σκέψεις και βεβαίως θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Ευχαριστώ. Η Φρανσέσκα Μπαλζάνη και εγώ εργαζόμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Συνεπώς δεν είναι η πρώτη μας συζήτηση για αυτό το θέμα. Και υποστηρίζω πλήρως αυτό που ελέγχθη σε σχέση με την ανάγκη στην Ευρώπη να έχουμε άτομα με καλύτερα προσόντα και δεξιότητες. Συμφωνούμε στην Επιτροπή με αυτή την ανάλυση όλοι. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Αυτό σημαίνει πρέπει να επενδύσουμε για τα παιδιά μας και για τους νέους ώστε να βρεθούν σε καλύτερη θέση σε σχέση με τα προσόντα τους να, να έχουν αναπτυχθεί καλύτερα. Όσον αφορά τώρα στο πολιτικό επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 έχουμε την αηφορία, την βιωσιμότητα, και έχουμε τα προγράμματα διαβίου εκμάθησης, το Εράσμους και ακόμη και τις νεολαίες τα προγράμματα συμβάλλουν πολύ προς αυτή την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε καλοί στην απόδοση, έχουμε καλή απόδοση δηλαδή, απορροφητικότητα και μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε και για τον επόμενο προϋπολογισμό και για το επόμενο MSF ότι όσα πράττουμε εδώ έχουν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Όλοι τώρα έχουν ξεκινήσει να συζητούν τι είναι η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και μπορούμε πολύ πιστικά να δείξουμε τι είναι. Είναι να προσεγγίζουμε τα άτομα, δεν πρόκειται για τα μεγάλα προγράμματα υποδομής, ασχολείται με ανθρώπους. Το Εράσμους, και η όλη προσπάθεια πλησιάσματος προς τον πολίτη της Ευρώπης. Πρέπει να τονίσουμε αυτό το επιχείρημα. Όσον αφορά τώρα το μέλλον των ανοιχτών κοινωνιών με πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτικές συνθέσεις, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το πολιτιστικό πρόγραμμα είναι να συμβάλλουμε προς, προς αυτόν τον στόχο. Ε, τώρα, ως προς την ανταγωνιστικότητα, τα προγράμματά μας πρέπει να αποτελούν μέρος της στρατηγικής, της ευρύτερης για, τον για την ανταγωνιστικότητα. Ανέφερα και την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας, Europeana και η χρηματοδότηση της Europeana πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέρος της στρατηγικής του 2020. Και όταν θα ασχοληθούμε με τον επόμενο προϋπολογισμό καθώς και με τον πιο μακρόχρονο σχεδιασμό πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφος συγγνώμη. Είπανε πολλοί συνάδελφοι πράγματα που ήθελα να πω, ιδίω η κυρία Τρούπελ. Ήθελα όμω να μείνω στο θέμα τη χρηματοδότηση του αθλητισμού. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητε χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα στον τομέα του αθλητισμού. Θα ήταν ίσω ε, αντιφατικό, ενώ έχουμε περισσότερε αρμοδιότητε, να έχουμε λιγότερα λεφτά ή σχεδόν καθόλου χρήματα. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν κάποιε προσπάθειε για να βρεθούμε στο ύψο, να αρθούμε στο ύψο αυτών των αρμοδιοτήτων ο πολιτισμός έχει πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά ο αθλητισμός όχι. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εισαγάγουμε και τον αθλητισμό σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αναφέρθηκε πάρα πολύ ο Έρασμος, που είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πιστεύω ότι τα προγράμματα Έρασμος έχουν κάνει περισσότερο για την ενότητα της Ευρώπης από ό,τι πολλές συνθήκες. Θα ήταν σημαντικό να τα διατηρήσουμε και όχι μόνο να τα διατηρήσουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να τα διευρύνουμε στο βαθμό του δυνατού. Επίσης, τώρα που έχουμε μια αυτόνομη εξωτερική πολιτική με πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεξιά και αριστερά, για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά και την πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω. Να δώσουμε μια υποστήριξη για να αναπτύξουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική για τα πολιτιστικά θέματα εναντί άλλων χωρών, άλλων υπήρων. <clears throat> σε πολλούς τομείς μπορούν να είναι πιο σημαντικοί και πιο αποτελεσματικοί άλλοι, ε, άλλες χώρες και άλλες ήπειροι, αλλά στην κουλτούρα δεν μας κερδίζει κανείς και πρέπει η Ευρώπη να το καταδείξει αυτό και να έχει την διαναπαραίτητη ακτινοβολία. Η κυρία Μπάντια Κουτσέτ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλτσάνη που ήρθε ενώπιόν μας για να μας εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπαλτσάνη Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτό το σχέδιο το οποίο θα μας δώσει η Κομισιόν, όπως είπε η κυρία Πάξ, στα τέλη Απριλίου και θα συζητήσουμε και ελπίζουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε επί τη βάση αυτού του σχεδίου. Αλλά για απόψε το απόγευμα έχουμε μια συνάντηση για την κατάρτιση, για τις νέες δεξιότητες και όλα αυτά, όπου ήμασταν παρόντες πολλοί από εμά. Η κυρία Πάκη είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ νόημα για τα θέματα που μας απασχολούν μας παρουσίασε πριν από λίγο η κυρία Πακ την κατάσταση που ήταν ρεαλιστική για να μην πω απεσιόδοξη, αλλά η κατάσταση βέβαια δεν είναι απλή, είναι αρκετά δύσκολη και δραματική. Και πρέπει, και φυσικά και εσείς πρέπει να μας βοηθήσετε, ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα πάντα. Αλλά η επένδυση στην παιδεία είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το θίξουμε. Δεν πρέπει να μειώσουμε την ε, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ακόμα και αν έχουμε ε, πίεση στο, στα δημοσιονομικά δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος να περικόψουμε τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειώσουμε λοιπόν αυτόν τον προπολογισμό. Πρέπει να λειτουργήσουμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη κατανομή πόρων. Δεν μπορούμε όμω να περικόψουμε τον προπολογισμό τη εκπαίδευση, γιατί αυτό θα είναι ένα τεράστιο πολιτικό λάθο κατά την άποψή μου. Μία ακόμα παρατήρηση. Σε σχέση με το ποσοστό της, ε, των προγραμμάτων ε, διαβίου εκπαίδευση που αφορά του ενήλικε το, την εκπαίδευση των ενηλίκων. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Μιλάμε για ένα 4%. Έχουμε όλο και περισσότερου ενήλικου σε ηλικία που εργάζονται. Έχουμε άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ανεργία, αλλά είναι άτομα τα οποία είναι <clears throat> ενήλικε. Χρειαζόμαστε αυτά τα προγράμματα να έχουν περισσότερου πόρους για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλα αυτά τα άτομα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την παιδεία του ενώ συγχρονώ συμμετέχουν στην κοινωνία μα με το να εργάζονται όχι σαν μία τάξη αδρανών ατόμων, αλλά σαν μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται. Η κοινωνία μα αλλάζει και πρέπει και εμεί να παρακολουθήσουμε αυτή την αλλαγή, να αλλάξουμε μαζί τη και να θεσπίσουμε του σωστού στόχου για να παρακολουθήσουμε αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ, Ρεκή Πρόεδρο. Η κυρία Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπαλτσάνη ιδίω, γιατί η μέθοδος στην οποία πρότεινε μου φαίνεται πάρα πολύ ε, θετική και αυτή η έγκαιρη παρουσία των επιτροπών θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα πιο θετικό διάλογο. Τρία σημεία θέλω να θίξω και να υπογραμμίσω. Πρώτον, συμφωνώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία ελέγξαν, αλλά πρέπει να τονίσω ακόμα ότι σήμερα <clears throat> πρέπει να έχουμε και μία συνειδητοποίηση ότι όλο το βάρος της κρίσης αυτή τη στιγμή βαραίνει τις νέες γενιάς. Αν δεν το λάβουμε αυτό υπόψη, δεν μπορούμε να εξισορροπήσουμε σωστά τον προϋπολογισμό μας και η Ευρώπη του 2020 στην οποία αναφέρθηκε πολύ σωστά η κυρία Μπαλτσάνη λόγω της στρατηγικής σημασίας και ακόμα και το ορόσημο του 2012 παίζει κάποιο ρόλο στο 2020 όταν έχουμε τέτοια στενότητα προϋπολογισμού εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ποιο θα είναι το σωστό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δώσουμε εμείς και να αναστρέψουμε την τάση στον προϋπολογισμό γιατί αυτό θα επηρεάσει και τα επερχόμενα έτη. Μιλάμε για την Ευρώπη 2020, την Ευρώπη των νέων δεξιοτήτων, <clears throat> της δυνατότητας να έχουμε μια συμμετοχή ως πολιτών το πιο ηλικιωμένων, μια πιο ευφυά μορφή κοινωνίας που θα περιλαμβάνει και τα πολιτιστικά θέματα. Μιλάμε για τον πάρα πολύ φιλόδοξο στόχο για τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε οι ελάχιστε συνθήκες για να υλοποιηθεί, να μπορούν όλοι οι νέοι στη ζωή τους να κάνουν σπουδές είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο είτε μέσα στα πλαίσια μιας εργασίας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και εδώ το πρόγραμμα Ερασμός, το οποίο είναι ένα από τα πιο επιτυχή προγράμματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτει ένα μικρό ποσοστό καταρχήν των νέων, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ να υπάρξει ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και των δυνατοτήτων εργασίας της. Πέραν του Εράσμου, του Ερασμού έχουμε και τον έρασμο για τους επιχειρηματίες και τον έρασμο για, για τους μαθητευομένους που εκεί πραγματικά η χρηματοδότηση είναι πραγματικά ανεπαρκέστατη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στο να έχουμε τη δυνατότητα για τους νέους να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Πέραν των θεμάτων του αθλητισμού που αναφέρθηκα, για τα οποία δεν υπάρχουν αρμοδιότητες, δεν υπήρχαν αρμοδιότητε και ω εκ τούτου δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθόλου χρήματα, υπάρχουν και νέα θέματα αρμοδιοτήτων όπω είναι ο τουρισμός. Δυστυχώ γίνεται μικροφωνισμό με κάποιο τηλέφωνο, με κάποιο κινητό τηλέφωνο. Υπάρχει ένα άλλο σημείο στο οποίο έχουμε θέσει μια προπαρασκευαστική δράση που είναι ο πολιτιστικό, η πολιτιστικός τουρισμός. Α, το μικρόφωνο μου είναι. Ζητώ συγγνώμη τους διερμηνείς και τα αυτιά τους. Ο πολιτιστικός λοιπόν τουρισμός και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την προώθηση του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι μια πολυθετική δράση που ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί και επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πέρα από την παιδεία υπάρχουν τα θέματα της, ε, του πολιτισμού. Μιλάμε για τους δημιουργικούς ε, πολιτιστικούς κλάδους, μιλάμε για το πρόγραμμα Media, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας βοηθάει να είμαστε ανταγωνιστικοί στον τομέα αυτό Ξέρω ότι η κυρία Πακ θέλησε να εξασφαλίσει ότι θα έχει τη σωστή χρηματοδότηση. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης μέσα στον χώρο ε, της, του πολιτισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνουν όλα αυτά τα κονδύλια που δίνονται για τα μέσα ενημέρωσης μόνο στο τωρινό επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλτσάνη για την παρέμβασή τη και ιδίω για τη μέθοδο την οποία έχει υιοθετήσει για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι πιο συνενετικό, πιο συμμετοχικό και που θα υποστηρίζεται από όλου. Ε, Συμμερίζομαι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για τη σημασία που έχουν μια σειρά από δράσει για του νέου, για τον αθλητισμό, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Απλώς θα ήθελα να κάνω κάποιες πολιτικές σκέψεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον προϋπολογισμό της και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει εδώ να δώσει μια, ένα μήνυμα ε, αντιστροφής κατεύθυνσης σε σχέση με τα εθνικά κράτη. Ενώ τα εθνικά κράτη περικόπτουν τα ποσά για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό θα ήταν θεμελιώδη. Για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και ενώπιον της κρίσης την οποία διατρέχουμε, να μπορέσει να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε <clears throat> μια τέτοια αντιμετώπιση. Αντίθετα, η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στι κατευθύνσει αυτέ για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ακόμα και αν τα κράτη-μέλη περιορίζουν τη χρηματοδότησή του. Να δείξει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να προχωρήσει στους τομείς αυτούς με θετικό τρόπο. Ένα άλλο στοιχείο είναι αυτό που έχει να κάνει με την Μεσόγειο. Σε μια στιγμή που έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση, υπογραμμίζεται από όλους το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει και στην νότια όχθη της Μεσογείου, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και εδώ δεν θα μπορούμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη αν δεν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει το αίσθημα ηθαγένειας και συμμετοχής στα κοινά θέματα στις κοινωνίες αυτές. Και εδώ πρέπει να δώσουμε υποστήριξη στα πολιτιστικά σχέδια, να υποστηρίξουμε προγράμματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν την κατάλληλη σχέση με την ευρωπαϊκή παιδεία και κουλτούρα, να υπάρξει και η επαφή των ε, νέων από την νότια όχθη της Μεσογείου με τους νέους από την βόρεια όχθη της Μεσογείου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει και ένα καινοτόμο ρόλο και είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε κάποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μπαλζάνη για την ε, έκθεση και θα ήθελα να αναφερθώ στα δημοσιονομικά προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προπολογισμό συρρυκνούτα σε πραγματικούς όρους κατά τη διάρκεια των δημοσιονομικών αυτών προοπτικών. Το 2007 δηλαδή ήταν περίπου το 1,3 του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τώρα ανέρχεται στο 1,12 μόλις του συνολικού ΑΕΠ. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια έχουν, ενώ έχουν διπλασιαστεί οι εθνικοί προπολογισμοί σε ονομαστικούς όρους τουλάχιστον, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό παρουσιάζει αύξηση μόνο κατά ένα τρίτο σε ονομαστικούς όρους. Αυτό δεν ε, αποτελεί καλό ιονό για το μέλλον. Και θα ήθελα να πω με την ευκαιρία αυτής της συνεδρίασης ότι θα μπορούσαμε με τα εφιστάμενα κονδύλια ήδη να δαπανίσουμε πιο ε, αποτελεσματικά τους πόρους μας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και τέτοιους τομείς προτεραιότητας. Θα ήταν καλό επίση στην Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο να μην δώσει αρνητικά μηνύματα στα κράτη-μέλη περιορίζοντας την ε, χρηματοδότηση σε στόχους που έχουμε ορίσει ως ε, επιδιοκτέους για, το, για τον ορίζοντα του 2020. Εάν περιοριστεί και άλλο προπολογισμό, να μπορέσουμε ε, από το 2015 και μετά να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Εάν θέλουμε περισσότερου ανθρώπου με υψηλή, επίπεδο μόρφωση, θα πρέπει ασφαλώ να ενισχύσουμε και τη χρηματοδότηση, τα κονδύλια για του νέου και τι σπουδέ του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε επίπεδα ισοδύναμα με αυτά των ΗΠΑ, τη Ιαπωνία και άλλων προηγουμένων χωρών. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω ότι θα πρέπει κάθε νέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει ότι έχει την ευκαιρία τουλάχιστον για ένα εξάμεινο να ε, υποφεληθεί του προγράμματος κινητικότητας στην εκπαίδευσή του, στην κατάρτισή του ε, μέχρι το 2020. Μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να είμαι απεσιόδειξος, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει, εφόσον μιλάμε για χρήματα, τουλάχιστον να ακουστεί αυτή η παρατήρηση. Ευχαριστώ κυρία Γάινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μπαρτσάνη ήρθε σήμερα το πρωί και στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου πάλι ζητήθηκαν περισσότερα κονδύλια για τις μεταφορές. Και θα πρέπει να ε, υπογραμμίσω ότι και τα θέματα βέβαια των, ε, του τουρισμού είναι σχετικά με τις μεταφορές, με την ευρία έννοια και κυρίως με τον τουρισμό και σε αυτό και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα έρασμου, σε παραδείγματα έχουν γεννήσει πολλέ προσδοκίε επίδο πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο αναπτύσσουμε διάφορε δραστηριότητε και εκδηλώσει, όπου προσπαθούμε να προσκαλέσουμε και αθλητέ και καλλιτέχνε και εκπροσώπου του πνεύματο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όμως με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε δεν μπορούμε στην πράξη να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε. Και μπορεί βέβαια να διακηρύσουμε ότι υποστηρίζουμε τον αθλητισμό, αλλά δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό. Και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα ε, οπτικής γωνίας και επιλογών προτεραιοτήτων. Γι' αυτό θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι είστε διατεθειμένοι να λάβετε υπόψη σοβαρά τις ανάγκες αυτών των συγκεκριμένων κλάδων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πακ, χωρίς μικρό το μικρόφωνο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μιλάμε ακόμα για τον προπολογισμό του 2012, στο πλαίσιο δηλαδή ακόμη των δημοσιονομικών, του δημοσιονομικού μας προγραμματισμού. Και θα πρέπει να ξέρουμε και ότι μπορούμε να δαπανίσουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε προβλέψει αυτή την πενταετία. Είχαμε προβλέψει αυτό, εκείνο και το άλλο για το κάθε πρόγραμμα, διάφορα ποσά τα οποία όμως είμαστε υποχρεωμένοι τώρα για τη φετινή χρονιά να περικόψουμε. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Προσπαθώ εδώ και χρόνια, αλλά δεν το έχω καταφέρει. Είναι δυνατόν να έχουμε ήδη λάβει μια απόφαση ότι θα πρέπει για κάθε χρόνο να υπάρχει το τάδε ποσό και μετά να πρέπει να το περικόψουμε. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι κονδύλια τα οποία αφιερώνουμε στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και που μπορούμε να αξιοποιήσουμε γι' αυτό που θα έλεγα κάπως ε, ρομαντικά ε, την ψυχή της Ευρώπης ή το μέλλον της Ευρώπης, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι α, κάτι περίσπιση θα το επιστρέψουμε στα κράτη-μέλη από τον προπολογισμό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε πάνω απ' όλα να εξαντλούμε κάθε δεκάρα που έχουμε στη θέση μας. Και το 12 θα είναι δύσκολο και το 13 θα είναι πιο δύσκολο ακόμα. Και επίσης. Δικά μα λεφτά εμεί δεν έχουμε. Μπορούμε να διαθέσουμε μόνο τα κονδύλια που μα δίνουν οι άλλοι. Φέρει πριν το πρόγραμμα για τα μέσα μαζική ενημέρωση, το Media, εάν αποφασιστεί ότι θα περικοπεί, ότι θα καταργηθεί κιόλα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε δεν το θέλουμε εμεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δυνατόν. Να μην ξέρουμε πώ λειτουργεί το πρόγραμμα, πόσα κονδύλια έχουμε, πόσα, τι μπορούμε να διαθέσουμε και να μην περνάει από το χέρι μα αυτό και μόνο οι κυβερνήσει να αποφασίσουν αν θα μα διαθέσουν τα κονδύλια. Φαντάζομαι ότι εσείς θα μας βοηθήσετε κυρία Μπαρτσάνη στον αγώνα αυτόν. Η Επιτροπή, ποιος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε όσα ελέγχθησαν, διότι συμφωνούμε με όσα υπόθηκαν. Και χαιρόμεθα για τις προτεραιότητες που προδιαγράφεται η εκπαίδευση. Πραγματικά έχει υψηλή προτεραιότητα. Τα περισσότερα προγράμματα που διαχειριζόμαστε συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Έχουμε 7 βασικά προγράμματα τα οποία συμβάλλουν ακριβώς στα 7 κέρια σημεία της στρατηγικής του 2020. Συνεπώς η διασύνδεση είναι πολύ σαφής. Όπως ελέγχθη από πολλούς, τα χρησιμοποιούμε τα χρήματα σωστά, χρησιμοποιούμε όλα επενδύοντας στην εκπαίδευση, στους ανθρώπους, στις ανταλλαγές, την απόκτηση δεξιοτήτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλωσορίζω όσα ελέγχθησαν και ελπίζω, όπως είπε η Πρόεδρος, ότι τουλάχιστον θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτά που αποφασίστηκαν μέσα στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε τα σχέδια που εξελισσόντουσαν τουλάχιστον να εφαρμοστούν πέρυσι με τη δικιά σας υποστήριξη και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ευρύτερα, μπορέσαμε να αποκτήσουμε πρόσθετα κονδύλια για τα περισσότερα προγραμματά μας. Χρειαζόμαστε να προσέξουμε τουλάχιστον για όλα τα προγράμματα για το 2012 να εξασφαλίσουμε τα ίδια κονδύλια, να μην υπάρξουν δηλαδή περικοπές σε σχέση με το φετινό έτος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Κυρία Μπαλτζάνη ξαναζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις όλους και όλες, από τις οποίες ε, <clears throat> εξέρχονται μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σας έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοναδικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το γεγονός ότι έχετε αρμοδιότητα για προγράμματα τα οποία έχουν λειτουργήσει θαυμάσια στο παρελθόν, όπως ε, υπενθύμησε η Πρόεδρο σας και όπως είπε και η κυρία Τρίπελ, είναι προγράμματα τα οποία έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες Ευρώπης και αυτό είναι κάτι το σημαντικό. <clears throat> για τους πόρους που αν τα συγκρίνουμε λοιπόν με τους πόρους που έχουν από τον προπολογισμό που δεν είναι περιορισμένοι, δείχνουν ότι έχουν μια τεράστια προσθέμενη αξία, γιατί έχουν άμεση επίπτωση για τους ανθρώπους και δημιουργούν αυτό το αίσθημα ότι ανήκουν σαν πολίτες στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Βέβαια, δεν είναι κάτι νέο το οποίο σας λέω, άμα σας πω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεγάλη πρόκληση γενναιών. Υπάρχει γύρω του πληθυσμού, αλλά πρέπει παράλληλα να δώσουμε μια πραγματική επένδυση για τους νέους. Οι νέοι χρειάζονται προσόντα για να μπορέσουν να συμμετέχουν και να είναι ανταγωνιστικοί σε έναν κόσμο ο οποίος ζητάει όλο και περισσότερα προσόντα. Και αυτό αφορά και τους ευνήλικες, γιατί ακόμα και αυτοί που δεν είναι τελείως νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσουν και να ανακατευθύνουν τις ικανότητές τους. Επομένως, <clears throat> το θέμα αυτό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της επένδυσης για τα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την ανακατεύθυνση των ικανοτήτων και των προσόντων είναι κεφαλαιώδες για το μέλλον μας. Πρέπει να είμαστε επίσης και συνεκτικοί με τον πρώτο στόχο της Στατηγικής Ευρώπης 2020. Περισσότερες θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας μεγαλύτερης ποιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Και επειδή 10 χρόνια μπορεί να φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι και πολύ μικρός ο χρόνος, αν σκεφτούμε τη φιλοδοξία του, των στόχων της Ευρώπης 2020, θα πρέπει να έχουμε μια συνεχή ε, επένδυση χωρίς να κάνουμε υπαναχωρήσεις για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Αναφέρθηκε επίση η ανάγκη, η αναγκαιότητα, ο προπολογισμό εν γέννη και οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουν και, συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα της λιτότητας που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι λοιπόν μια άλλη μορφή του να σκεφτόμαστε να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική γωνία και πιστεύω ότι εδώ ο πιο σημαντικός στόχος τον οποίο θα πρέπει να τονίσουμε θέτοντας την ε, φιλοδοξία της Ευρώπης 2020 στα πλαίσια του προϋπολογισμού είναι να έχουμε κάποιες προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να επενδύουμε με τρόπο μόνιμο και σταθερό και να αφήνουμε σε σχέση με αυτές τελείως κατά μέρος τα επιχειρήματα της κρίσης και της ανάγκης περιστολής των δημοσίων πόρων. Πρέπει λοιπόν να είναι η τομή συνευραλική σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και που θα δίνουν και μια σωστή κατεύθυνση για τα κράτη-μέλη και μια μόνιμη αντιμετώπιση. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι θέλουμε να τα σπρώξουμε προς την κατεύθυνση μιας πιο μακρόπνοη στρατηγικής που πολλές φορές λόγω της κρίσης, της συγκυρίας και των πολιτικών που πολλές φορές αλλάζουν όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις είναι πολύ πιο δύσκολο τα κράτη-μέλη να την διατηρήσουν. Και αυτό οδηγεί σε μεγάλες ζημίες πολλές φορές για τους ίδιου πολίτε. Μιλήσαμε επίση και για τις νέε αρμοδιότητε, για τον αθλητισμό, για τον τουρισμό, για τα θέματα της Μεσογείου. <clears throat> Νομίζω ότι όταν να έχουμε πόρους για τις νέε αυτέ αρμοδιότητε, αυτό είναι προβληματικό, όπως είναι προβληματικό το να έχουμε πόρους για την στρατηγική του 2020 το ο προπολογισμό αυτό του 2012 και ο επόμενος προϋπολογισμός, η επόμενη προπολογισμό μέχρι το 2020 θα απαιτήσουν μια συνεκτικότητα σε επίπεδο θεσμικό μεταξύ των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια πραγματικά θεσμική αξιόπιστη πολιτική θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σειρά από προτεραιότητες οι οποίες θα είναι λειτουργικές αλλά για τις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα δώσουμε την απαραίτητη δημοσιονομική υποστήριξη. Αυτό είναι το έργο λοιπόν στο οποίο πρέπει να αποδειθούμε όλοι μαζί με μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για τις αρμοδιότητες που έχουν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ, να καταλήξουμε σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι συνεκτικός με τις στρατηγικές που έχει θεσπίσει για τον εαυτό της Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουμε εμείς ψηφίσει ως Κοινοβούλιο και στις πρόσφατες Ολομέλες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων που θα είναι η οδηγή για τις επιλογές μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα πρέπει <clears throat> σιγά σιγά μέσα στις επιμέρους επιτροπές να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε όλες αυτές τις προτεραιότητες που θα δώσουν συνεκτικότητα στις επιλογές μας σε όλες τις φάσεις και αυτό περιλαμβάνει και τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και φυσικά θα οδηγήσει στην κατάθεση τροπολογιών που είναι η πιο δύσκολη και λεπτή μορφή ε, φάση του προπολογισμού. Ευχαριστούμε κυρία Μπαλτσάνη. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και σε εσά και στον εαυτό μας. Και αρκετά λεφτά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Πάλι για λεφτά μιλάμε δηλαδή. Πρόκειται για το νέο. Ναι, ναι, όλα, όλα, όλα από τα λεφτά περιστρέφονται. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό λοιπόν το οποίο θα, υπάρχει από το, θα, έπρεπε να, θα πρέπει να υπάρχει από το 2013 και επέκεινα και είχαμε δημιουργήσει πέρσι μια επιτροπή η οποία εργάζεται ήδη εδώ και ένα χρόνο για να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες μας για το μέλλον ώστε να μπορούμε να είμαστε ισχυροί στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Ε, και έχουμε ένα μέλος μας στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, ο οποίος είναι ο κύριος ε, Ιβαν, στον οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τι έχει γίνει σε αυτή την Επιτροπή, γιατί σύντομα θα τελειώσει η θητή αυτής τη επιτροπή, και η εντολή τη. Παρακαλώ κύριε Ιβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, μιλάμε για τα χρήματα που θα έχουμε στη διάθεσή μας μετά το 2014, δηλαδή μιλάμε για τα χρήματα που θα χρειαστούμε και τα οποία δεν θα τα έχουμε μετά το 2014. Το πρόβλημα με αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μοιάζει να επιμικίνεται και μέσα στο επόμενο πολιετές Συζητάμε πολλά οριζόντια θέματα τα οποία πρέπει να επικυρώσουμε εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη δικιά μας αρμοδιότητα. Όσον αφορά τα οριζόντια θέματα, η διάρκεια και η ευκαμψία αυτού του πλαισίου και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αυτά είναι τα βασικά. Όσον αφορά τη δομή και την ευκαμψία του μελλοντικού πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, η ευκαμψία ειδικότερα, ή για να το πω διαφορετικά, όσο πιο εξειδικευμένο είναι ένα κεφάλαιο, όσα περισσότερα υποκεφάλαια έχει, τόσο λιγότερο εύκαμπτος είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή δεν μπορούμε να μεταφέρουμε από το ένα, το ένα κονδύλι ένα κονδύλι από τη μία στην άλλη θέση. Από μία γραμμή του προϋπολογισμού σε μια άλλη. Η Κομισιό υπέβαλε δύο προτάσεις. Η μία ε, έχει τρία κεφάλαια, το οποίο μας δίνει μεγάλη ευκαμψία. Όμως έχει το μειονέκτημα ο προϋπολογισμός να είναι πιο δύσκολος στην εποπτεία του. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση που αφορά την στρατηγική 2020 με τρία κεφάλαια και τέσσερα τμήματα. Σας έλεγα ότι αυτή η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι λιγότερο εύκαμπτη, διότι έχουμε τα τέσσερα υποκεφάλαια, τα οποία κατακαιρματίζουν, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό για την επόμενη περίοδο. Όσον αφορά τώρα τη διάρκεια, το που έχει σημασία είναι η αξιοπιστία. Η πολιτική και η δημοσιονομική. Όσο μακρύτερη διάρκεια, τόσο, καλ, τόσο λίγο... Τόσο, ε, τόσο περισσότερο έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμάσουμε μακροχρόνια προγράμματα σε διάφορους τομείς. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν για ένα πενταετές και η Επιτροπή Σούρε πιστεύει ότι αυτό το πενταετές πρέπει να αντιστοιχεί με την εντολή του Κοινοβουλίου. Μου μοιάζει υπερβολική αυτή η πρόταση, διότι αυτοί που θα σχεδιάσουν το δημοσιονομικό πλαίσιο για πέντε χρόνια δεν είναι αυτοί που θα το υλοποιήσουν, για την προετοιμασία πριν πολύ χρόνο και αν θέλετε οι βουλευτές θα φτιάξουν το σχέδιο για τους επόμενους βουλευτές. Δεν έχει νόημα αυτό. Ε, τώρα, ένα πλαίσιο δεκαετές με σημαντική ανασκόπηση στη μέση, με δυνατότητα μεταρρυθμιστική, ένα τέτοιο, μια τέτοια διάρκεια δέκα ετών μας δίνει δυνατότητα προβλεψιμότητας και υπάρχει και η συμβιβαστική λύση, η επταετής, είναι το πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ αυτή τη πρόταση, δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν συνηθίσει το επταετές, η κατάσταση λειτουργική αρκετά καλά και μια μεταβολή δεν θα ήταν χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε άλλους τομείς μπορούμε να μιλήσουμε για την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Για την Επιτροπή Πολιτισμού δεν αμφισβητείται διότι και τα προγράμματα παιδείας, πολιτισμού, σπορ, και για τα μίντια είναι προγράμματα που έχουν καταδείξει τη χρησιμότητά τους. Δηλαδή συνενώνουμε κονδύλια και αυτό δίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα προγράμματα. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι όσον αφορά τη στρατηγική του 2020 υπάρχουν δύο στόχοι που συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση. Πρέπει να μειώσουμε κατά 10% τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο και πρέπει να ενισχύσουμε τα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης. Οπωσδήποτε, συνεπώς, η παιδεία είναι μια προτεραιότητα. Ε, αναφέρομαι βεβαίως και στη διαβίου μάθηση και στους, ε, ε, στα προγράμματα για τους πολίτες της Ευρώπης η έκθεση λοιπόν θα συζητηθεί αύριο, πρόκειται για την Επιτροπή Σούρε, και δυστυχώς δεν καλύπτονται τα πράγματα πολύ καλά για την περίοδο μετά το 2014, διότι όσο σημαντικές και αν είναι οι προτεραιότητες, δεν υπάρχουν κονδύλια μετά το 2014 και αύριο θα συζητήσουμε και την έκθεση Καποντήλια για τους δημοσιονομικούς πόρους. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Πακ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την έκθεση του κυρίου Μάλλον περιμένουμε την έκθεση στην γνωμοδότηση του κυρίου Ιβαν ε, για την Επιτροπή για την Κρίση, τη ΣΟΥΡΕ. Έχουμε και τον άνθρωπο εργασίας και αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις τροπολογίες μπορείτε να καταθέσετε έως τις 22 Μαρτίου στις 12 του μεσημέρι. Πρόκειται για μια έκθεση που βλέπετε στην ημερήσια διάταξη επόμενη συνεδρία τον Απρίλιο για ψηφοφορία. Ο κύριο Μάτουλα έχει στον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια, όχι μόνο για την έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ, αλλά και σε, σχέδιο, και σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου. Συνολικά, θα έλεγα ότι συμμερίζομαι τους στόχους που αναφέρονται. Και επιτρέψτε μου, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κεφάλαιο για την στρατηγική της Ευρώπης το 2020. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με 7 ετή διάρκεια είναι η καλύτερη επιλογή με μια αναθεώρηση στη μέση της περίοδου. Νομίζω ότι αυτή η διάρκεια ήδη έχει δοκιμαστεί αποτελεσματικά. Η ευκαμψία είναι εξίσου σημαντική, δηλαδή θέλουμε λιγότερες δημοσιονομικές γραμμές, απλούστευση και ευκαμψία για το σύνολο του προϋπολογισμού. Τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Συνεπώς, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι τα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας είναι πραγματικά υποδείγματα, μοντέλα σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή είναι ιστορίες επιτυχίας, ορα, ε, ορατότητας μεγίστης. Και αν μιλάμε για μεταβολές θα πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε η επιτυχία που έχουμε καταφέρει να μην χαθεί μελλοντικά. Οπωσδήποτε όταν μιλάμε για την απλούστευση των δημοσιονομικών γραμμών το το συζητούμε, διότι θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε κανδύλια με μεγαλύτερη ευκολία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε πρώτα τα κονδύλια τα διαθέσιμα, εφόσον ενδεχομένως δεν υπάρχει δυνατότητα να τα αυξήσουμε. Δηλαδή μελλοντικά με τι πρόκειται να πραγματικά να λειτουργήσουμε. Μεγάλο ερώτημα. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και εθνικής. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να έχουν αναμφισβήτητα την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία <coughs> εκ του γεγονότος ότι λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι θα έχουμε τα μέσα να, να εξασφαλίσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα τρίγωνο. Νεολαία, σπορ και απασχόληση. Από τη μία πλευρά δεν πρέπει να ξεχνούμε το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο στην κατηγορία των νέων. Μιλάμε από την άλλη πλευρά για διαβίου μάθηση. Ωραία. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου όλους αυτούς τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο και οι οποίοι Απλώς έρχονται να προσθεθούν στον τεράστιο αριθμό των ανέργων. Όταν μιλάμε για νέες αρμοδιότητες, δεν πρέπει να ξεχνούμε και το σπορ. Έχω κατά νου τη μαζική άθληση. Δεν ε, σημαίνει αυτό ότι ε, δεν θέλω τον πρωταθλητισμό, αλλά με ενδιαφέρει ο μαζικός αθλητισμός και κυρίως ο αθλητισμός των νέων ίσως θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα το στόχο μας και να μειώσουμε το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου α, μέσω του αθλητισμού, μέσω των σπορ. Και χάρη στα σπορ ίσως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την υγεία των συμπολιτών μας, διότι συχνά ξεχνάμε την παχυσαρκία. Οι ενήλικες δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες, διότι τα προγράμματά μας ήταν ορατά, ήταν μια πραγματική επιτυχία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν ακόμη περισσότερο. Οπωσδήποτε είναι γνωστά αυτά τα προγράμματα, διότι βλέπουμε ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι πάρα πολύ υψηλό. Αλλά όσο περισσότερο τα συζητούμε, τόσο περισσότερο θα καταλάβουν και οι άλλοι ότι δεν είναι λογικό τα 7 βασικά μας προγράμματα να μειώνονται σε χρηματοδότηση από μία χρονιά σε άλλη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τρίβιλ, ευχαριστώ πολύ Θα ήθελα για μια φορά να αναφερθώ στην ε, πολιτική αντιπαράθεση ε, που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε από τα κράτη που, είναι, που εισφέρουν καθαρά στον προπολογισμό με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμα για πάγωμα των ποσών για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι τομείς που μα απασχολούν θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλε δυσκολίε. Αυτή η σκληρή γραμμή όμως μπορεί, εάν δεν περάσει, να έχει να αφήσει ως συνέπεια ε, περιορισμούς ως προς την ανάπτυξη των ποσών για το θέμα τα ακριβώς αυτά. Δηλαδή να μην έχουμε ε, παρά μόνο μια πολιτική λιτότητα σε αυτούς τους τομείς. Άρα θα πρέπει αν θέλουμε να ενισχύσουμε τα κονδύλια για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, θα πρέπει από κάπου αλλού να τα αντλήσουμε τα κονδύλια. Και ξέρουμε τι αντιπαραθέσει και μέσα στι πολιτικέ μα ομάδε μεταξύ αρθρωτική πολιτική, περιβαλλοντική, πολιτισμού, εξωτερική. Όμω, και το έχω επισημάνει πολλέ φορέ, πρέπει, πρέπει πλέον να δώσουμε μια σαφή γραμμή για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Όπου έχουμε εμεί πολύ σημαντικά επιχειρήματα να προωθήσουμε τι δικέ μα επιλογέ. και κυρίως χάρη και στον άνθρωπο του συναδέλφου μπορούμε να δώσουμε και ποσοστά με τα ποσοστά εφαρμογής και επιτυχίας του βαθμού στον οποίο μπορούμε χάρη στην πολιτική αυτή να πλησιάσουμε και να αγγίξουμε τον Ευρωπαίο πολίτη και έτσι να βελτιώσουμε την αποδοχή από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κάποια θέματα λοιπόν διαρθρωτικού χαρακτήρα σχέση με τις πολιτικές αυτές επιλογές. Φερρυπίν, πρώτα απ' όλα, ε, χρονικό πλαίσιο 5-7 ή 5 συν χρόνια. Τα 7 χρόνια είναι η περίοδο η επταετία είναι η περίοδος στην οποία ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, η οποία με βρίσκει αρκετά σύμφωνη, διότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματισμού, ενώ τα 5 συν 5 σαν πλεονέκτημα θα επέτρεπαν βέβαια να υπάρχει μια αναθεώρηση και αξιολόγηση ότι έχουμε καταφέρει, χωρίς να χρειάζεται από την αρχή να τα αναθεωρήσουμε όλα και να τα ξανασυζητήσουμε. Εάν όμως η κατάσταση όσον αφορά τις επιλογές αυτή τη στιγμή είναι μάλλον δυσμενής για τις δικές μας θέσεις, είναι ρεαλιστικά και πραγματικά και ε, ε, πολιτικά ορθή η επιλογή του να πούμε ότι δεσμεύουμε αυτές τις επιλογές τα επόμενα δέκα χρόνια ενώ ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη στην προσεχή ε, πενταετία του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε πάντα να έχουμε υπόψη σαν πολιτική σκοπιμότητα και βέβαια σε αντιπαράθεση με το ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστό. Ο κύριο Κέλλη χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο και πάλι ο κύριο Κέλλη. Πολλά από τα οποία ελέγχθησαν σε σχέση με το 2012 έχουν να κάνουν με τις νέες αρμοδιότητες του αθλητισμού και του τουρισμού. Και πραγματικά πρέπει να ρωτήσει κανείς τι νόημα έχει να έχει κανείς πρόσθετες αρμοδιότητες αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε προγράμματα στον τομέα αυτό. Αυτό πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, στεναρά το τόνισε ο Μάρκο και η Χέλεν. Και πέραν του θέματος λογικής, έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι στα θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, αλλά από πλευράς ε, από πλευρά τουρισμού και αθλητισμού έχουμε τεράστιο δυναμικό να αναπτύξουμε περισσότερο δραστηριότητε και αρμοδιότητε σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να το πράξουμε και να το κάνουμε τμήμα των προτάσεων μα σχετικά. Για το 5 συν 5 ή για το 7, τα 7 χρόνια για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, εγώ θα ήθελα να ακούσω τα επιχειρήματα αυτών οι οποίοι μίλησαν για 5 χρόνια για να καταλάβω γιατί. Εγώ νομίζω ότι 7 χρόνια είναι μια πιο πρόσφορη αντιμετώπιση. Αν υπάρχουν όμως αντιμαχόμενα επιχειρήματα, θα ήθελα να ακούσω αυτή την αντιμετώπιση. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι 5 συν 5 ή θα είναι 7, αν θα έχουμε διάμεση ε, αναθεώρηση. Όλα αυτά πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διαρθρωμένης συζήτησης και επιχειρηματολογίας. Η κυρία Σενάλοβα για να κλείσουμε. Χωρίς μικρόφωνο. Σμόλκοβα. Σμόλκοβα λέει η κυρία Σενάλοβα. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις προ... τα όσα είπαν οι συνάδελφοι οι οποίοι υποστηρίζουν την ε, πενταετία ως λύση, την επταετία συγγνώμη ως λύση. Ε, ωστόσο θα ήθελα και περισσότερη ευελιξία στην έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες. Είναι καλό βέβαια το μέσον ε, και αποτελεσματικό προκειμένου να ε, αντλήσουμε κορδίλια, αλλά μπορεί να υπάρχουν και πολλές καταχρήσεις. με τόση μεγάλη ευελιξία ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε από τα κράτη-μέλη κατάχρηση ε, που τελικά θα οδηγήσει στα μη επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σας ένα παράδειγμα από ένα επεισόδιο που είδαμε πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Πρώην Επίτροπος ο πρώην επίτροπο για την Εκπαίδευση, ο κ. Φιγγέλ, ήρθε στις Βρυξέλλε για να ζητήσει μεταφορά ποσών από τον τομέα της εκπαίδευση του πολιτισμού και της απασχόλησης σε προγράμματα για τις μεταφορές. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι οι μεταφορέ είναι σημαντικός τομέα. Οι υποδομές της μεταφορέ, αλλά θα έπρεπε από αλλού να χρηματοδοτούνται και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εναλλακτικέ πηγέ, ενώ για την εκπαίδευση δεν είναι εύκολο να βρεθούν εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Οι πέντε στόχοι της στρατηγικής του 2020, ασφαλώς δεν θα έχετε αντίρρηση, είναι στόχοι με ε, προτεραιότητα την εκπαίδευση ή απαιτείται η εκπαίδευση για να ε, εξυπηρετηθούν, να ικανοποιηθούν. Το να μην επενδύσουμε στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό σημαίνει από τώρα να αποφασίσουμε ότι δεν θα ικανοποιήσουμε αυτού του στόχου του 2020. Και γι' αυτό νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε το στο δημοσιονομικό πλαίσιο και το επίπεδο τη ευελιξία, θα αντιμετωπίσουμε αρκετέ δυσκολίε, Θα είναι δύσκολο να μεταφέρουμε και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μεταφερθούν ε, άλλα κονδύλια από την εκπαίδευση προ άλλου τομεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σμόλκοβα, διορθώνει λοιπόν η πρόεδρο. Έχουμε τελειώσει αυτή τη συζήτηση. Μήπω θέλει η Κομισιόν να μα πει κάτι. Παρακαλώ. Uh, uh, Απλώς να σας υπογραμμίσω ότι είναι απίθανο να υπάρξουν πρόσθετα ποσά, οπότε πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες. Έχουμε πολύ καλά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό και την παιδεία, αλλά πρέπει να διακριβώσουμε από πού θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολο από ότι είναι στην πραγματικότητα, γιατί ακόμα και αν είναι σημαντικός για ορισμένου ο προπολογισμό μας, είναι σε συνολικό επίπεδο τα θέματα πολιτισμού και παιδείας λιγότερο από το 2% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακόμα και μια σημαντική αύξηση του προπολογισμού μας δεν είναι σημαντική αύξηση συγκρινόμενη με το συνολικό ύψος του προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε κάποιους συναδέλφους μας να παραιτηθούν από κάποια χρήματα, αλλά σε απόλυτους όρους δεν μιλάμε για τεράστια ποσά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Επίσης, αν θέλουμε να έχουμε πρόσθετα κονδύλια, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταδείξουμε ότι παίρνουμε τα πράγματα σοβαρά, ότι δαπανάμε με επωφελή τρόπο τα χρήματα αυτά, ότι κοιτάζουμε με κριτικό πνεύμα αυτά που κάνουμε για να δούμε αν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα σε πιο επιτυχείς δράσεις, να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερα τα προγράμματά μας. Το κάνουμε λοιπόν αυτό με πολύ μεγάλη φροντίδα γιατί ξέρουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση της αίτησής μας για χρήματα αν είμαστε και εμείς αυτοκριτικοί. Νομίζω ότι αυτά τα οποία ελέγχθησαν είναι λίγο τρομακτικά, πιστεύω για μένα, ότι στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονται χρήματα για τις ελιές. 2,5 δισεκατομμύρια για ελιές όχι, συγγνώμη, 2,5% δεν είναι, δεν Κάτι κατάλαβα, δεν κατάλαβα καλά. 2,5% του προϋπολογισμού. Και εμεί έχουμε 1,8% για τα μέσα ενημέρωσης, για την παιδεία, για την νεότητα, για την συμμετοχή των πολιτών. Λοιπόν, ίσως λοιπόν με αυτά τα στοιχεία μπορεί κανείς να δείξει την παραλογή το παράλογο αυτού του θέματος. Τώρα εγώ σαν Γερμανίδα τι ξέρω για τις ελιέ, δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αλλά ίσως μπορούμε να πάρουμε λίγο από τις ελιέ να δώσουμε στι πατάτε ή κάτι τέτοιο. Μια επανεξισορρόπηση. Πάντα στη γεωργία υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπορεί να βρει κανεί. Κύριε Ιβάν, θέλετε να πείτε κάτι. Η κυρία Σμόλκοβα ήθελε να πει κάτι ακόμα. Μάλλον να της εξηγήσουμε πώς θα λειτουργήσει το θέμα της ευελιξίας, το 5 συν 5. Μπορείτε να της εξηγήσετε καλύτερα για το θέμα των ε, χρονικών διαρκειών. Ως προς τη διάρκεια της ε, δεκαετίας, 5 5 χρόνια δηλαδή, Πρόκειται για τη διάρκεια για την, οποία, περίοδο για την οποία εκφράστηκε η μεγαλύτερη υποστήριξη για τα προγράμματά μας. Πρόκειται για την περίοδο δηλαδή μετά το 2014. Και στην περίοδο αυτή θα πρέπει τα προγράμματα που τώρα είναι εξελίξει να αναθεωρηθούν για να τροποποιηθούν. Τόσο λοιπόν και οι διαδικασίε του ελέγχου τη επιτήρησης εφαρμογή των προγραμμάτων ή τη εποπτεία του τρόπου με τον οποίο του ελέγχου του τρόπου με τον οποίο δαπανήθηκαν τα ποσά θα υφίστανται, θα ε, υπάγονται στις νέες διαδικασίες. Και θα... Είναι σκόπο να μην χρειαστεί να αρχίσουμε από το μηδέν, να μην χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τα πάντα. Βέβαια κάθε στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά η πενταετία, και γι' αυτό το λόγο η πενταετία δεν αρκεί. Γι' αυτό προτιμώ τα 10 χρόνια, 5 συν 5, που μπορεί όμως για κάποιους να φανούν υπερβολικά μακρά περίοδος. Γι' αυτό και έχει σημασία η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, εις βάθος. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε εις βάθος και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι 10 χρόνια ακούγεται πολύ, αλλά αν το δούμε ως 5 συν 5 με ενδιάμεση αναθεώρηση εις βάθος, διατηρούμε και την ευελιξία μας, αλλά και την δυνατότητα για την επιβολή ε, τροποποιήσεων εκεί όπου κάτι δεν έχει πάει καλά. Ευχαριστώ πολύ. 22 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12 προθεσμία για κατάσταση των υπολογιών πάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης με τον κύριο Κέλλη, ο οποίος ασχολείται με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια συνολική προσέγγιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. την γνωμοδότησή μας την έχει αναλάβει εκ μέρου μα την έχει αναλάβει ο κύριο Κέλλη, στον οποίο δίνω το λόγο για το σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας πολιτικός τομέα για την Επιτροπή μας, διότι ασχολείται και με την εκπαίδευση και με την παιδεία και με την νεολαία και τον πολιτισμό. Το Νοέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε μια ανακοίνωση της Κομισιόν όσον αφορά μια συνεκτική προσέγγιση για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΑΕ. ΕΕ. Και έτσι ανοίγει η συζήτηση. Έχουμε ένα πλαίσιο εν ώψη της ε, γρήγορης ε, τεχνολογικής εξέλιξης λόγω της ε, τεχνολογίας cloud και για λόγους διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η πρώτη προστατευτική οδηγία εμφανίστηκε το 1995 και προσπάθησε να βρει ισορροπία ανάμεσα στην κυκλοφορία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Στη συνέχεια είχαμε άλλες οδηγίες που κάλυψαν τις εξελίξεις στον ηλεκτρονικό τομέα. Τώρα ερχόμαστε στο άρθρο 8 που δίνει νέα νομική βάση για την προστασία ανθρωπίνων ατομικών δικαιωμάτων. Online και offline. Αυτό επιτρέπει στους ε, νομοθέτες να δώσουν μια νέα νομική προστασία. Υπάρχουν οι τέσσερις τομείς στους οποίους αναφέρθηκα. Δηλαδή θέλουμε προστασία, θέλουμε διαφάνεια, προστασία των ανηλίκων, των ανηλίκων και ενίσχυση της συνειδητοποίησης και της ενημέρωσης. Δηλαδή από τις κυβερνήσεις και από τους παρόχους υπηρεσιών ε, κοινή ωφελία, πρέπει οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τη διαχείριση των πληροφοριών. Η προσβασιμότητα βεβαίω είναι θέμα κλειδί και με απλά λόγια οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα όταν έχουν ε, ε, θέματα προστασίας παιδιών. Η Κομισιόν πιστεύει λοιπόν ότι οι διατάξεις του 1995 δεν είναι αρκετά σαφείς και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησής μου, επειδή ακριβώς τα θέματα άπτονται στην νεολαία και στην παιδεία, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε να προσδιορίσουμε τα δικαιώματα και τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και των δύο μερών. Αυτό είναι το κλειδί και τα δύο μέρη έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και αυτό ε, έχει ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά. Δεν θέλουμε δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών μας να διαρρεύσουν προς τρίτους. Οι ελεγκτές των δεδομένων δεν πρέπει να έχουν ιδιοκτησία των δεδομένων επάπειρο. Αυτό είναι ένα άλλο κλειδί, δηλαδή η πληροφορία δεν πρέπει να γίνει ιδιοκτησία τους επάπειρων. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκπαίδευση συνειδητοποίηση εκ μέρους των πολιτών. Η γρήγορη μετα... τεχνολογική μεταβολή σημαίνει ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα της ενημέρωσης. Και για τα άτομα και προς τους πολίτες δηλαδή και προς τους ελεγκτές των δεδομένων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, τη σχετική νομοθεσία δηλαδή. Καμιά φορά οι πληροφορίες βρέθηκαν σε λάθος χέρια χάνοντας ας πούμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα λάπτοπ, καταλήγουν τα δεδομένα εκεί που δεν είναι προς συμφέρον κανενός. Το προσωπικό ε, ακόμη στις δημόσιες αρχές πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις τους. Και τα άτομα, ιδιαίτερα οι νέοι, και αυτοί χρειάζονται εκπαίδευση για να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, τις ευθύνες τους ιδιαίτερα σε σχέση με το υλικό που βάζουν σε ιστοσελίδες, στα κοινωνικά δίκτυα επίσης, διότι όλα αυτά μπορούν να μείνουν ίσως για πάντα και να είναι επιζήμια για τα ίδια τα άτομα που τα ανήρτησαν αργότερα όταν θα αναζητούν εργασία. Όλα αυτά είναι πρόσφατες εξελίξεις και χρειαζόμαστε νομοθετική ρύθμιση και χρειαζόμαστε ακόμη και συνειδητοποίηση των κινδύνων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και η σχετική εκπαίδευση. Επανέρχομαι και λέω ότι χρειαζόμαστε να έχουμε εκπαιδευτικό κομμάτι και κομμάτι συνειδητοποίησης. Υπάρχουν διάφορες άλλες πτυχές που θα ήθελα να αναφέρω και αρχικά είχα περιλάβει το δικαίωμα να μπορεί κανείς να ξεχαστεί αλλά δεν, μπορούσα, δεν είχα αρκετό χώρο για να βάλω όλες τις ιδέες μέσα. Ακόμη πρόσφατα είχα, είχα κάποιες επικοινωνίες σε σχέση με το άρθρο 9 που αναφέρεται στη δημοσιογραφία. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω να έχω τα σχόλια των συναδέλφων και τις τροπολογίες τους. Και σίγουρα μαζί θα μπορέσουμε να περάσουμε ένα σημαντικό μήνυμα προς την Κομισιόν σε σχέση με τις προτεραιότητες μας σε συνάρτηση με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για φέτος. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία και θα ήθελα δυστυχώς να σας πω ότι κυρία Πρόεδρε δεν μπορέσω να είμαι εδώ αύριο για την εθνική μας γιορτή και θα γιορτάσουμε την ημέρα του Αγίου Πατρικίου με μπύρα και προς τιμήν σα μπορώ να πιω κι άλλη μια-δυο εμπειρίε, αν αυτό σας αρέσει. Πολύ ευχαριστώ, Η κυρία Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον ε, Τζον Κέλλη για, για το σχέδιο γνωμοδότηση για να υποχρεώσω το εξή ξεκινώντα ότι η προστασία τη νεολαία σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και τις νέες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες και κυρίως να σκεφτούμε τι θα κάνουμε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα τα δίκτυα κοινωνική δικτύωση, τα social networks, πώς θα πλησιάσουμε σε αυτόν τους νέους. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί ε, να φέρουν ως επιπτώσεις ε, αυτά τα ε, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης που δεν γνωρίζουν ως, ίσως ε, τις συνέπειες τους οι δηλαδή όταν στέλνουν φερειπίνα την εικόνα ενός λουλουδιού ε, ως ευχετήρια κάρτα μέσα από το διαδίκτυο, ίσως δεν έχουν καν συνείδηση του πόσα και ποια προσωπικά του στοιχεία μεταδίδονται. Και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να ε, ε, γνωρίζουμε και πώς ακριβώς μπορεί να γίνει ότι μάλλον δεν υπάρχει ακριβής γνώση για το πώς, ε, τι χειρισμοί γίνονται μέσα από αυτό το διαδίκτυο και την κοινωνική δικτύωση. Πολλές φορές ε, υποτίθεται ότι απευθυνόμαστε σε νέους, αλλά τελικά πρόκειται για ηλικιωμένου, ότι δεν γράφει κανεί πάντα παράτητα τη σωστή του ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ευκαιρίε για συνάντηση, για επικοινωνία, αυτέ που προσφέρει το ίντερνετ, αλλά το δικαίωμα τη το δικαίωμα του να μπορεί κανείς να διαγράψει όποτε θέλει, ανα πάσα στιγμή και απόλυτα τα δεδομένα του από τη βάση δεδομένων μιας ε, ενός ε, κοινωνικού δικτύου είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ <clears throat> και εγώ μπορώ να συνεχίσω ε, μετά από αυτά που είπε και η προλαλή σας. Θα θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Κέλλη και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης. Σε κάποια σημεία όμως πρέπει να είναι πιο έντονο το περιεχόμενο αυτό, να το τονίσουμε περισσότερο. Πιστεύω πάντα ότι η καλύτερη μορφή προστασίας των νέων είναι η αρμοδιότητα και ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης. Εμεί θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέσα ενημέρωσης, έναντι αυτών που θεωρούν ότι ήδη υπάρχει αρκετός έλεγχος στα κράτη-μέλη. Γιατί και τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο στα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ζητήσουμε να αναλάβουν αυτά τα θέματα και τα θέματα της εκπαίδευσης σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και όχι απλώς να τους λέμε πόσο σημαντικά είναι. Πρέπει τα παιδιά ήδη από την παιδική τους ηλικία να μάθουν πώς θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα νέα μέσα ενημέρωσης ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτά τα μέσα και να ξέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ίντερνετ και να αποφύγουν τις σχολείους ατραπούς. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη του πάροχου υπηρεσιών γιατί αυτή είναι Εξάλλου αυτοί οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα προσωπικά για όλους μας. Δεν πρόκειται μονάχα για τους νέους. Εμείς θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε τι στοιχεία κατακρατάει ο πάροχος υπηρεσιών για μας και σε ποιο βαθμό αυτά τα δεδομένα μπορεί να περάσουν σε τρίτους. Δεν είναι μονάχα το θέμα λοιπόν της παράδοσης στοιχείων που είναι υποχρεωμένοι να κρατούν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά να υπάρχει η υποχρέωση του κάθε ενός να ελέγξει ότι τα στοιχεία τα προσωπικά τα οποία δεν θέλουμε να κρατάει ο πάροχος για μας να μπορούμε να τα σβήσουμε οριστικά. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε έμφαση σε αυτό το σημείο και όχι απλώς να τονίσουμε αυτό το σημείο αλλά να κάνουμε την απέτηση, να διατυπώσουμε την απέτηση να γίνει κάτι τέτοιο ώστε να υπάρξει πραγματικά μια υποχρεωτική εκστρατεία για την ενημέρωση και την εκπαίδευση από παιδική ηλικία μέχρι και τους ενήλικες σε σχέση με τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Κυρία Χάνιμπαου. Äh, ξεκινώ με αυτά που είπε η κυρία Κάμερη προηγουμένω νομίζω ότι είναι ένα επίμαχο θέμα ακόμα και στη δική μου πολιτική ομάδα το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πάροχους υπηρεσιών. Το αν πρέπει να υπάρχει ρύθμιση ή όχι. Υπάρχουν δύο σχολές. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση και μείωση των ελευθεριών. Άλλοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν κανόνες για να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλους. Και εγώ ανήκω σε αυτό το δεύτερο στρατόπεδο. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα πώς θα πρέπει να το πράξουμε αυτό τις ρυθμίσεις και ποια είναι τα όρια τα οποία θα, στα οποία θα πρέπει να φτάσει αυτή η ρύθμιση. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί μονάχα στο θέμα αυτό της ε, αντιμετώπισης των παρόχων υπηρεσιών. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει καταρχήν αυτονομία σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης για τους νέους για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν με έναν τρόπο ο, ο οποίος θα είναι επωφελής. Και εδώ πρέπει να υπάρξει και ένα στοιχείο αυτορύθμισης. Και τώρα στα λέω στα αγγλικά για τον κύριο Κέλλη. Κάνατε την ε, πρόταση, το σημείο 6, η προστασία δεδομένων για τα παιδιά και τους ανήλικους. Δεν κατάλαβα ακριβώ εγώ ίσως, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς να, αναφέρετε εδώ ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στα κοινωνικά δίκτυα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους ανήλικους. Δεν κατάλαβα ακριβώς πού ήταν η πρότασή σας, αν θέλετε να δείτε τον αντίκτυπο σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ηλικία ή όχι. Μια ερώτηση για τον κύριο Κέλλη, αλλά θα να κάνω πρώτα μια προκατακτική παρατήρηση. Έχω ζήσει για μεγάλο μέρος της ζωής μου σε μια χώρα όπου πολλά ήταν απαγορευμένα και όπου οι πάντες ήξεραν τα πάντα. Ζω τώρα σε μια χώρα όπου υπάρχουν ελάχιστε απαγορεύσει, ή δεν απαγορεύεται τίποτα σχεδόν. Και ναι, κάποιο μπορεί να γνωρίζει κάποιο προσωπικό δεδομένο, κάποιο όχι. Θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν τι επιφυλάξει μου απέναντι σε κάθε μορφή απαγόρευση. Επίσης, από την εμπειρία μου βλέπω ότι είναι πολύ πιο ασφαλής νομικά η προστασία όσο πιο ε, έντονη είναι η νομική παρέμβαση υπέρ της προστασίας των παιδιών, τόσο πιο αναποτελεσματική είναι. Αυτό βλέπω και από την πατρίδα μου. Είναι λιγότερο αποτελεσματικές οι απαγορεύσεις που εισάγονται με τον νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πράξουμε και θα ήθελα να υποστηρίξω ρητά τι προσπάθειε του κυρίου Κέλλη και την προσέγγιση του. Αλλά με απασχολεί το εξής ερώτημα. Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ γρήγορα. Και όποιο έχει παιδιά στην ηλικία που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το ίντερνετ, ασφαλώ έχει διαπιστώσει είναι πολύ πιο εύκολο για αυτά να ε, βρούνε λύσεις και να προσαρμοστούν ε, στην τεχνολογία του υπολογιστή από ότι ένας ανήλικας. Άρα θα ήταν καλό να τα οθήσουμε προς μια πιο δυναμική προσέγγιση αυτής της τεχνολογίας. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο στην έκθεση να σημειώσουμε ότι πρέπει αυτή η διαδικασία να είναι να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώ επαναρχόμαστε στον ε, κύκλο, στον επαναλαμβανόμενο κύκλο, ότι τα παιδιά μαθαίνουν πολύ γρήγορα κτλ. κτλ. Η κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Κέλλη για αυτή την έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον, που κάνει πολύ σωστέ επισημάνσει. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ρύθμιση του διαδικτύου και ξέρω ότι είναι ευρύτατο θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, όμως δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση πουθενά, καμία επικοινωνία οποιοδήποτε τύπου που να, να μην έχει κάποια αρρύθμιση. Η απαγόρευση ίσως είναι μια σκληρή λέξη. Όμως κάπου πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο σε σχέση με το τι είναι αποδεκτό και τι απαράδεκτο. Περί αυτού πρόκειται άλλωστε συζητήσαμε σε αυτή την Επιτροπή τις φρικτές εικόνες των παιδιών που εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Είναι παράνομες αυτές οι εικόνες στα κράτη-μέλη, αλλά δεν θα ήταν πολύ καλύτερο αν δεν μπορούσαν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μου. Ε, δηλαδή υπάρχει ανάγκη για προστασία ε, για ορισμένους χρήστες. πρέπει να τους προστατεύσουμε από τη βλάβη την οποία θέλουν να επιφέρουν άλλοι. Συνεπώς, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε προστασία των δεδομένων και υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση. Τώρα υπάρχουν και λιγότερο σαβαρά ζητήματα βεβαίως, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί. Βεβαίως η εκπαίδευση on media θα βοηθούσε στην καταπολέμηση ε, και αυτό θα ήταν χρήσιμο και για τους γονείς και για τα παιδιά. Δηλαδή, ε, οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν τι μπορούν να βλέπουν ε, τα παιδιά στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ. Το να είναι γνώστης της χρήσης των μέσων ενημέρωσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά ακόμα και από τον εαυτό τους. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πάντα ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπορούν να προστατευτούν αν δεν ξέρουν από, την, από νεαρή ηλικία ποια είναι, τα επικοινά σημεία. Πρέπει όμως να έχουμε και κάποιους εκπαιδευτές, κάποιους δασκάλους που να καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε αυτούς που θα διδάξουν στα παιδιά. Γιατί και αυτοί θα πρέπει να γνωρίσουν τις τεχνικές αυτές που πολλές φορές ξέρουν, την ξέρουν λιγότερο αυτή την τεχνολογία από ότι οι μαθητές τους. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σε αυτό το τομέα και να εξασφαλίσουμε ότι οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί θα αντιμετωπίσουν αυτή την προβληματική για να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα προστατευτούν από παιχνίδια τα οποία μπορεί να έχουν ένα πολύ επικίνδυνο χαρακτήρα. Έχετε το λόγο και πάλι. Είναι πάρα πολύ σύντομα σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Τρίπελ. Για να μην υπάρξει μια παρεξήγηση, θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τους παρόχους να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των χρηστών ή αυτών που παρέχουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί να αναλάβει όλη την ευθύνη για αυτά τα πράγματα ο πάροχος. <clears throat> Ένα δεύτερο πρόβλημα για την προστασία των νέων έχουμε το πρόβλημα ότι ουσιαστικά κυνηγάμε τους ανεμόμυλους όπως ο Δον Κιχώτης. <clears throat> Μιλάμε πολλές φορές για όρια ηλικίας για τους νέους. Λέμε, ξέρω εγώ, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ορισμένα είδη περιεχομένου στην ε, τηλεόραση μετά από πριν από μια ορισμένη ώρα ή στο οτιδήποτε τέτοιο, αλλά πολλέ φορέ οι γονείς αφήνουν τα παιδιά του να κάθονται και να βλέπουν νυχτερινά προγράμματα στο, στην τηλεόραση χωρί να προστατεύουν τα παιδιά του Και δεν του νοιάζει ότι κοιτάνε τα παιδιά τους, δεν κοιτάνε στην τηλεόραση. Υπάρχει πάντα λοιπόν μια θεά περιοχή όπου πρέπει να δώσουμε βοήθεια για να αποφευθούν ορισμένα πράγματα, αλλά με την επίγνωση ότι οι τελικοί αποδέκτες αυτών των ε, μέτρων θα πρέπει και αυτοί να παίξουν το δικό τους ρόλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντα υπάρχει στην προστασία των νέων και πρέπει να υπάρχει και η συνένεση των γονέων και των ίδιων των νέων για να προστατευτούν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στη συζήτηση με τα σχόλιά τους. Βεβαίως είναι πολύ λεπτός, ευαίσθητος αυτός ο τομέας περισσότεροι σχολίασαν αφενός την ανάγκη να υπάρχει επαρκής ελευθερία για να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους το διαδίκτυο, αλλά αναφέρθηκαν επίσης και στην προστασία ειδικότερα των νέων. Το θέμα είναι μέχρι ποιου σημείου προστασία. Ο κύριος Μπίσκι έχει δίκιο. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με το διαδίκτυο και θα βρουν ε, τρόπους να, να ξεπεράσουν οποιαδήποτε απαγόρευση θα βάλετε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να νομοθετήσουμε. Ε, δημιουργείται την ευκταία κατάσταση η οποία ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένη ηλικία κτλ. Μιλάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρείται ένα υλικό το οποίο δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο για άτομα κάτω των 15, αλλά πρέπει να υπάρχει σχετική νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων. Είναι ζωτικό αυτό. Ειδικότερα αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αν βάλουν κάτι στο διαδίκτυο να αποφύγουν να μπορεί να διαγραφεί αυτό ε, αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το εξασφαλίσουμε γιατί στο κάτω-κάτω την ευθύνη βεβαίω την έχουν οι χρήστες αλλά και ο πάροχος έχει σοβαρή ευθύνη καθώς και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Έχετε πολύ δίκιο πρόεδρε όταν λέτε ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους εκπαιδευτικούς διότι τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με όλους αυτούς τους μηχανισμούς από ότι οι δάσκαλοι τους. Οι νέοι μετά γίνονται δάσκαλοι βέβαια πολλοί από αυτούς. Πρέπει να δημιουργήσουμε την πιο ισόρροπη κατάσταση. Αυτό είναι το ευκταίο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν τροπολογίες από τους συναδέλφους και ότι ο κύριος Σκέλη θα τις δει με χαρά. Έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες μας τη Δευτέρα στις 21 Μαρτίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Άρα, ας βιαστούμε. Σημείο 6. Έχουμε διαγράψει από την ημέρη σε διάταξη. Και τώρα, και κλεισμένο των θυρών, η συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παρόντες και παρακαλώ όποιος δεν έχει δουλειά στη συνεδρίασή μας να αποχωρήσει και οι προσκεκλημένοι βέβαια. Να μείνουν μόνο οι συντονιστές και το προσωπικό τους.